So you read yours and then. Right, ladies and gentlemen, dear colleagues, please be seated. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Πάλι έχουμε αργήσει, αφού προσπαθήσαμε κάπως να προλάβουμε όσο μπορούσαμε στη διάρκεια του γεύματος. Πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί με το χρόνο από την πλευρά της Επιτροπής ΑΦΕΤ. περιμένουμε τον Κροάτι Υπουργό και τον ε, ε, Πρόεδρο του ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν σας καλωσορίζω στην κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Περνάμε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν σχόλια εγκρίνεται αυτή. Τα πρακτικά από τις 6 Νοεμβρίου 2019 νομίζω να εγκριθούν. Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις εγκρίνονται και αυτά. Και να καλωσορίσω τα μέλη της ΔΕΒΕ και ιδίως τον πρόεδρο της ΔΕΒΕ, τον κύριο Τομπέ που κάθεται δίπλα μου Έχουμε τώρα επενημέρωση από την Επιτροπή ΑΦΕΤ και στο δεύτερο γύρο δημοτεύσεων με το Συμβούλιο για το θέμα του ε, εργαλείου για την διεθνή συνεργασία. Ε, στις διαπραγματεύσεις που είδε πάλι ο κύριος Τομπέ έχει ε, μοιραστεί το κείμενο της ε, με τις τέσσερις στήλε και από τις 19 Σεπτεμβρίου έχουμε το σχετικό κείμενο που μοιράστηκε για τον πρώτο τρίλογο ε, από τις 12 μάλλον Δεκεμβρίου και για την δυνατότητα της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέσο για νέο ανάπτυξης και νέο συνεργασίας. Ε, Παρακαλώ τους εισηγητές να μας τα πούνε από τη δική τους πλευρά. Ευχαριστώ, Ντέιβιτ, και χαίρομαι που βλέπω ότι σιγά-σιγά προχωρούμε. Προχωρούμε επί της ουσίας της πρότασης για το εργαλείο προενταξιακής βοήθειας, διεθνούς μάλλον συνεργασίας. Ευχαριστώ τους εισηγητές για την μέχρι τώρα συνεργασία τους και όπως είπες θα πρέπει τώρα να δούμε τι πρόοδος έχει επιτελεστεί για ουσιώδη ζητήματα πριν τις τελευταίες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για, για, το, διεθνές, ε, για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και ιδίω για τους συγκεκριμένους στόχους μας. Τα οικονομικά στοιχεία κυρίως όπως έχει οριστεί σε οριζόντιο επίπεδο και από τους δικούς μας εισηγητές Ελπίζουμε ότι το, ο προγραμματισμός για τις καταπήκουσε ανάγκες από την Επιτροπή θα ξεκινήσει το δυνατόν συντομότερα, ώστε να παραταθούν τα ισχύοντα προγράμματα πέραν του 2020. Αυτό θα ελαφρύνει την πίεση να κλείσει συμφωνία ε, με κάθε τίμημα. Και ανταυτού, μόνο εφόσον χρειαστεί, θα υπάρξουν κατεπήγοντα μέτρα για να πάμε προς ένα τελικό μέσο που είναι καταλληλότερο και αποτελεσματικό μέσα στο μεταβαλλόμενο διεθνές ε, σκηνικό και προκειμένου να ε, βασιστούμε και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε ένα εργαλείο που να βασίζεται στις φιλοδοξίες μας με πραγματικό κοινοβουλευτικό έλεγχο και ε, προσδοκίες. Εδώ να δώσω το λόγο στους εισηγητές για το θέμα αυτό. Παρακαλώ, David, να ξεκινήσουμε με το ε, μέσο διεθνούς ε, συνεργασίας. Ποιος θέλει το λόγο για τη γειτονία, ανάπτυξη και διεθνή συνεργασία. Δεν είναι εδώ οι εισηγητές. Κάποιος πρέπει να λάβει το λόγο όμως. Γκάλερ, Αρενά, Γκέρενς, Γιετσουβιτσιένε. Ναι, αλλά δεν ήμουν ε, στην συνεδρίαση της Επιτροπής ε, και του Τριλόγου, οπότε ήθελα να ευχαριστήσω τους εισηγητές. Είχαμε την συνεδρίαση προετοιμασίας πριν από κάθε γύρο τριμερών διαλόγων και οι συνομιλίε με τους σκιώδεις εισηγητές καθώς και τους εισηγητές των Επιτροπών Μπάτ και Θάμ, ήταν πολύ αποτελεσματικές. Ελπίζω να συνεχίσουμε με αυτό το επικοδομητικό πνεύμα και να, συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε σε αυτό το τόσο περίπλοκο ντοσχέ. Και επίση θα πρέπει να υπάρξει και, συνεργασία για το, και η ανάλογη συνεργασία και για το εργαλείο πενταξιακή βοήθεια 3. Ελπίζω ότι οι επόμενοι εισηγητέ τα ίδια θα πούν και ότι θα συνεχίσουμε αποτελεσματικά με τον επόμενο τριμερή διάλογο στις 20 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελε κάποιο άλλο να προσθέσει κάτι. Μάλιστα, πρόκειται για ένα μηχανισμό που είναι σημαντικός εφόσον ε, συγκεντρώνει όλα, όλους τους ε, μηχανισμούς με βάση την κύρια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε λοιπόν μια ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου μας σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης αυτής. Είναι σημαντικό να μείνουμε ενωμένοι σε αυτή τη δύσκολη διαπραγμάτευση μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου. Έχουμε τον πρώτο τριμερή διάλογο και συμφωνήσαμε στη μεθοδολογία με μια ομάδα που προετοιμάζει τις τεχνικές αποφάσεις και ευχαριστώ όλους όσοι εργάζονται εκεί και από πλευρά ε, πολιτικών ομάδων και από πλευρά γραμματεία, γιατί είναι πολύ δύσκολο το καθήκον που έχει αναλάβει, χρειάζεται πολύ χρόνο ε, και υπομονή και του ευχαριστώ. Χάρη σε αυτή την τεχνική προσπάθεια, ε, καταφέραμε να πάμε πιο εύκολα, αν θέλετε, στον τριμερή διάλογο για να μπορούμε να πάρουμε αποφάσει που δεν θα μπορούσαν να ληφθούν αν δεν είχαμε το τεχνικό σκέλο έτοιμο βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τρία μη ίσονο σημασία, θα έλεγα, προβλήματα αυτή τη στιγμή που ακόμα εκκρεμούν. Το πρώτο αφορά τον ρόλο των τοπικών αρχών. Θεωρούμε σημαντικό πλευρά θέση του Κοινοβουλίου να δώσουμε έναν ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρηματοδότηση τη εξωτερική πολιτική. Δεν είναι μία θέση την οποία συμμερίζεται όμω το, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, πρέπει να συνεχίσουμε να περασπιζόμαστε αυτή τη θέση. Όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στο επίπεδο των ε, πολιτών, τόσο πιο αποτελεσματικό θα είναι αυτός ο μηχανισμός. Το δεύτερο σημείο που δημιούργησε δυσκολίες είναι ότι η πολιτική προτεραιότητα θα πρέπει να περάσει από το πλαίσιο του rapid response, άμεσης ανταπόκρισης ε, που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάλι για το Κοινοβούλιο είναι θεμελιώδης σημασία να μην πάμε προς τα εκεί, γιατί στην άμεση ανταπόκριση δεν υπάρχει προγραμματισμός. Όμως σε νέους μηχανισμούς όπως είναι αυτοί εδώ οι δύο, ε, εμείς θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερο ρόλο ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσο περισσότερο πηγαίνουμε λοιπόν προς την άμεση ανταπόκριση, τόσο λιγότερο θα εμπλεκόμαστε εμείς ως Κοινοβούλιο. Και τέλος, θέλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο συνδέεται με τις ε, χώρες της Αφρικής, Καραϊβικής ε, και του Ειρηνικού. Υπάρχει μια γεωγραφική προσέγγιση όπου διακρίνουμε την Αφρική από τις υπόλοιπε ε, περιοχές. Όμως η Κοτονού βασίζεται στην ευρύτερη περιοχή Καραϊβικής και Αφρικής για σημαντικές προκλήσεις και εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή την προσέγγιση για αυτή την ε, πολιτική ομάδα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία συζήτηση αυτή τη στιγμή που εκκρεμούν. Βέβαια, μέχρι να τα συμφωνήσουμε όλα, δεν έχουμε συμφωνήσει τίποτα, έτσι ισχύει πάντα. Θα συνεχίσουμε να τα εξετάζουμε λοιπόν στις ε, διάφορες ε, ομάδες τεχνικής βοήθειας και τριμερού διαλόγου. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιος άλλος θα ήθελε να πάρει τον λόγο. Από την ΤΕΒΕ, μάλιστα. Προσπαθώ να βάλω μια σειρά. Γιατί πρέπει να κλείσει αυτό το θέμα σε πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Όσο ασυνησυγήτρια αυτή τη σημαντική έκθεση, θα ήθελα να μιλήσω για τα εκκρεμή ζητήματα. Το πλαίσιο πολιτική. Έχουμε συμφωνήσει επί τη πλειονότητα ε, των διατάξεων αυτού του άρθρου, όμω υπάρχουν ακόμα κάποιε διαφωνίε ό,τι αφορά τον ορισμό των ε, δευτερογενών πόρων ε, πολιτική καθοδήγηση. Ομάδα εργασία, επίπεδο επιτροπή Συμφωνήσαμε να το, να το αφήσουμε ανοιχτό αυτό το ζήτημα και να κλείσει όταν θα έχουμε συζητήσει τη συνολική διακυβέρνηση του μηχανισμού. Δεύτερον, συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών. Στο άρθρο για τις Γενικές Αρχές, το Συμβούλιο ζήτησε την, ε, να προσθεθεί ε, και ο όρος ε, συμφωνία, σύνδεσης ή ελεύθερων συναλλαγών σε διάφορες διμερείς συμφωνίες, εταιρικής σχέσης και την υλοποίησή τους. Στη δική μας πρώτη ανάγνωση δεν υπάρχει καμία αναφορά σε εμπορικές συμφωνίες. Συνεχίζονται συζητήσεις στην ομάδα του Κοινοβουλίου για το πώς θα το χειριστούμε. Και τέλος, ε, οι πρωτοβουλίες με ηγετικό ρόλο της Ένωσης. Η εντολή μας συμπεριλαμβάνει την διαγραφή της ε, παραγράφου αυτή στο άρθρο 15 που μιλάει για τη διαχείριση προκλήσεων και προτεραιοτήτων που προβλέπει ε, την ανταπόκριση σε νέες πρωτοβουλίες ε, των οποίων ηγείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα θέλαμε ως Κοινοβούλιο να διατηρήσουμε αυτή τη ε, διάταξη. Η συζήτηση αυτή προβλέπεται υπό το πακέτο διακυβέρνησης εφόσον η Επιτροπή συνδέει αυτή τη συζήτηση με τις άλλες διαδικασίες για το λεγόμενο μαξιλαράκι που είναι ένα επιπλέον και μεγάλο αποθεματικό ευέλικτης χρήσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Γκέρνς δεν είναι εδώ. Δύο συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο. Γκονζάλε και Ντεμορέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνω βέβαια ότι στο στάδιο του τριμερούς διαλόγου που βρισκόμαστε δεν έχουμε προχωρήσει σε συγκεκριμένα ζητήματα. Εγώ όμως θέλω να κάνω έκκληση στους εισηγητές, όπως και τους κοιόδης εισηγητές, για να μην ε, ξεχάσουν το δρόμο που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα για τη συνεργασία τη μεταβατική. Αναφέρομαι στο 5% για τη συνεργασία και τις χώρες μέσου εισοδήματο. Η συνεργασία αυτή δεν πρέπει να μειωθεί γιατί θα αποτελούσε οπισθοδρόμηση σε σχέση με τόσα έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Και επιπλέον θα κινδυνεύαμε αν επικεντρωθούμε ε, σε μία ήπειρο μόνο την Αφρική για την ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία βεβαίως τη θέλουμε, αλλά να ξεχνούσαμε τη Λατινική Αμερική, αυτό δεν θα ήταν σωστό. Η συνεργασία με τη Λατινική Αμερική πρέπει να συνεχιστεί και να συνεχιστεί όπως κάνουμε και τώρα, που είμαστε οι πρώτοι στη συνεργασία αυτή. Ευχαριστώ πολύ πάντως και ελπίζω να το αυτό οι συγητές και οι σκιώδεις συγητές. Ευχαριστούμε κυρία Κοντζάλες. Μορέλ. Εκτός μικροφώνου. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε για τις διαπραγματεύσεις και τη Γραμματεία για τη συστηματική ενημέρωση. Πολύ σύντομα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θέλουμε αποτελεσματική και διαφανή διαπραγμάτευση και τα σχετικά εργαλεία για τη διεθνή συνεργασία, την εξωτερική πολιτική και την αναπτυξιακή να είναι ε, αποτελεσματικά. Έχουμε ήδη πει ότι για τη διεθνή συνεργασία χρειάζονται κονδύλια για την ανάπτυξη που όμως να ε, χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτική εκπαίδευση ενδεχομένως και στην Αφρική να μην χρησιμοποιούνται για την ε, απομάκρυνση των μεταναστών παρόλα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε στη σωστή κατεύθυνση, εκεί όπου έχουμε ήδη ξεκινήσει να οδεύουμε και επίσης θα χρειαστεί πολύ περισσότερη διαφάνεια με, την, ε, ε, με τον συντονισμό των διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων και διαφανέστερες διαδικασίες για την αναπτυξιακή πολιτική όπως ζητούν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις από τις οποίες λαμβάνονται κονδύλια. Αυτό είναι και το μόνο σημείο επίκριση. Ευχαριστώ, συνάδελφε. άλλε παρεμβάσεις. Ωραία, λοιπόν. Περνάμε στο 15 ε, ο λόγος τους συνεισηγητές στο εργαλείο προενταξιακής βοήθειας, το IPA3, για να μας ενημερώσουν για την εξέλιξη των δημοτεύσεων. Συνεισηγητές είναι ο κύριο Πίτσουλα και η κυρία Σόφκου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Στις 12 Δεκεμβρίου είχαμε τις αρχικές συνομιλίες με την Φιλανδική Προεδρία ε, και για τους κανόνες για το μέλλον του εργαλείου πενταξιακής βοήθειας. Παρά τους πολλούς τομείς σύγκλησης θα πρέπει να δούμε τις ε, διαφορές απόψεως απόψεων σε πολλά σημεία του ντοσιέ. Ο κύριος Πίτσουλα και εγώ έχουμε καταρτήσει ε, έναντι του Συμβουλίου της Προτεραιότητας του ε, Κοινοβουλίου για τη στρατηγική χρηματοδότηση στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον. Έχουμε επιμείνει ότι χρειάζεται η απαραίτητη χρηματοδότηση, αλλά μπορεί να πηγαίνει μαζί με την ενισχυμένη λογοδοσία και δημοκρατική ρεσιμότητα και να υπάρξουν μηχανισμοί για την πλήρη ή ε, και αμερόληπτη αναστολή του μηχανισμού εφόσον χρειαστεί. Θα πρέπει να υπάρξει προβολή επίση τη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, γιατί με καλύτερη στόχευση των προσπαθειών επικοινωνία μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεράστια δουλειά που έχει γίνει ευρωπαϊκή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στι χώρε ένταξη. Να ολοκληρώσω λέγοντα ότι τεχνική δουλειά μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων για το κείμενο του Εργαλείου προταξική Βοήθεια 3 συνεχίζεται. Οι διαπραγματεύσει θα εξαρτηθούν από τι λεπτομέρειε στην ε, χάραξη των, των μηχανισμού του εργαλείου αυτού. Κύριο Σπίτσουλα, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά είχαμε πολύ καλέ αρχικέ διαπραγματεύσει με τη Φιλανδική Προεδρία ε, και πέραν των προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου που ανέφερε η κυρία Σόφκο, επιμείναμε στα βασικά θέματα τη διαθέσμική φύση τη συνεργασία και του ρόλου του Κοινοβουλίου για να θέσουμε τι σωστέ προτεραιότητε για την προενταξιακή χρηματοδότηση. Παροτρύναμε το Συμβούλιο να επιταχύνει συνολικά τα σημεία ε, του διαμαρτυρικού κειμένου που βρίσκονται εντό αγγελών. και να προχωρήσουμε σε ένα πλήρω νομοθετικό κείμενο. Δυστυχώ, η οριζόντιες ε, διατάξεις που έχει επιβάλει αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο δυσκολεύουν την έβρεση συμβαστικών λύσεων για πολιτικά ζητήματα και δεν μπορεί έτσι να κλείσει το όλο θέμα. Επιμείναμε ότι η εντολή του Ευρωκοινοβουλίου για τις κατεξοδότηση πράξεις προβλέπει οι κατεξοδότηση αυτές πράξεις να χρησιμοποιούνται και για την επικαιροποίηση των παρατημάτων ε, των κανονισμών και για να μπορούν να γίνουν σωστές επιλογές στρατηγικού προγραμματισμού. Όπως ανέφερε ήδη ο Πρόεδρος κατά τη διάρκεια των Ευρωπαϊκή, παροτρύναμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει ένα πρόγραμμα κατ' επίξω ανάγκη στα πλαίσια του πολιτισμού συνομικού πλαισίου ω προπόθεση για να προχωρήσουμε. Θα πρέπει όλα αυτά να μπορούν να λειτουργήσουν από την 1η Ιανουαρίου 2021. Ευχαριστούμε τον Νίνα, ευχαριστούμε Γέλενα Σόφκο. Ε, σχόλια από την πλευρά σας, ερωτήσεις, συμβουλές. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Τόμας, κάτι από την πλευρά σου. Ευχαριστώ, όλους τους συναδέλφους για όλες τις δηλώσεις τους. Τις ερχόμενες εβδομάδες θα έχουμε ίσως περισσότερα να πούμε. Πολύ καλή τελική αυτή φράση. Ολοκληρώνουμε την ενημέρωση από του συνεισηγητέ για τα δύο κοινά θέματα ΑΡΦΕΤ-ΔΕΒ ή τέλο πάντων τη διαδικασία τριμερού διαλόγου τη ΑΦΕΤ. Εύχομαι στου συναδέλφου καλό υπόλοιπον ημέρα και